τις ψηφοφορίες τώρα. Η πρώτη μας ψηφοφορία αφορά τη σύσταση ε, επιτροπής, ε, επιτροπής για τις εκπομπές ε, ε, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Κύριος Κάρβερ. Nope. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφε, με ακούτε. Είναι ασύνηθες. Πολύ ασύνηθες. Η πρόταση που θα ψηφίσουμε. Ανακοινώθηκε μόλις 7 το βράδυ χτες, εδώ. Όταν είχαμε μια δράκα συναδέλφων παρούσα. Είναι κανονικό αυτό. Διότι έπρεπε αντιρρήσει, ενστάσεις και σχόλια να γνωστοποιηθούν πριν τι 8 το βράδυ στο Προεδρείο. Και είχαμε μια φούχτα μονάχα βουλευτές παρόντες. Αυτό ήταν μη δημοκρατικό, αντιδημοκρατικό και παράξενο. Εντάξει, καλώς. Σας ενημερώνω ότι ταυτόχρονα έβγαινε και ε, στο διαδίκτυο και μπορούσατε να έχετε ενημερωθεί. Okay. Εντάξει, προχωρούμε ψηφοφορία για την ελόγω επιτροπή. Είναι ονομαστική η κλίση, αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Trecem ακόμα προχωρούμε στην επόμενη ψηφοφορία για τον Ιμπραήμ Χαλάουα. Ε, ε, έχουμε ένα κοινό ψήφισμα. Σημείο 5. Πρόεδρε, απλώς ήθελα να δεχτεί το κοινοβούλιο ότι Ιμπραήμ Χαλάουι, οι δύο αδελφές του είναι εδώ, για να δουν ομόφωνη υποστήριξη ελπίζουμε για απελευθέρωση του αδελφού τους Ιμπραμ Χαλάουι. Καλωσορίζουμε λοιπόν τις αδελφές του εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και προχωρούμε λοιπόν στην παράγραφο 5 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε και ε, ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά. Άρχη ψηφοφορία πέρας. Εγκρίνεται. Felicitări. Συγχαρητήρια. Το επόμενο θέμα, η κατάσταση της Μαλδίβες. Έχουμε ένα κοινό ψήφισμα από διάφορες πολιτικές ομάδες. Τροπολογία 2 ψηφιπέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σημείο 11 παράγραφος αρχίζει ψηφοφορία ονομαστικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 1 είπε Κατά. Αποχές. απορρίφθηκε. Το σύνολο του ψηφίσματος ε, ε, ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία, Μαλαισία. Κοινή πρόταση ψηφίσματος διαφόρων πολιτικών ομάδων. Έχουμε την τροπολογία παρελθόν 3, ψηφιπέ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 12, όχι. Μα ήταν προφανές το αποτέλεσμα. Παράγραφος 12. Αρχίζει η ψηφοφορία, ονομαστικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Η παράγραφο 2, ψηφιπέ. Συγγνώμη, τροπολογία 2 κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 14. Το αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Adoptat εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμένα είπε κατά, αποχές, απορρίψεται. Το σύνολο του ψηφίσματος είπε κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έχουμε τώρα την έκθεση της κυρίας Καλνιέτε Αρχίζει η ψηφοφορία. Μία ενιαία πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Λόχ Μπίλερ. η ψηφοφορία. Μία πάλι ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερη έκθεση Λόχ Μπίλερ. Έχουμε την τροπολογία παριθμών 1 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμών 4 ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 Η τροπολογία παριθμό 3. ψήφιπε Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 33. ψήφιπε Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμό 5. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η αιτιολογική σκέψη I σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα με ονομαστική κλίση αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στη πρόταση ψηφίσματο ολοκληρώνοντα την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η τροπολογία παριθμών 17D. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 5 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 18D υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμών 6 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασ. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 2 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 22 με ονομαστική κλίση αρχής υποφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 23 αρχίζει ψηφοφορία. Ένας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 26 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 27. Αρχίζει η ψηφοφορία. Votul λιέστε εγκείς. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 28 με ονομαστική κλίση αρχίζει η ψηφοφορία λήξης απορρίπτεται η τροπολογία 29 ψηφιπέ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 30 άρχιτη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται τροπολογία 31 άρχιτη ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 32 αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 33. αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34, έχει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35, ονομαστική κλίση και πάλι, έχει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 36, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμό 2 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 7 με ονομαστική κλίση αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 37. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38D τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 δι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση αρχής ψηφοφορία τώρα πέρας απορρίπτεται η 14 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 υπέ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 4 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα Votul este închis. Ε, πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα το σύνολο του ψηφίσματος ηλεκτρονικά, α, όχι, ε, απλά Είπε. κατά, αποχές, εγκρίνεται. It was obvious. Είναι σαφές το αποτέλεσμα. Η έκθεση του κυρίου Πρέντα τώρα ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο. Εμποτρίβα. Υπέρ κατά, λέει ο πρόεδρος, και αποχές και εγκρίνεται έξι χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το 7. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο υπέρ. Δε, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίε. Και εγκρίνεται. 22. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 27. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Χωριστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 37. Χωριστική ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Punctul 46 cade. 54. 46 στο αρχικό κείμενο ε, ψηφίσαμε πάνω στο 54 χωρίς ψηφορία το πρώτο υπέρ. Ψηφίζουμε. πέρασε Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56. Χωριστή ψηφοφορία. Ονομαστική. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απολύτω. 65. Αυτή η ψηφοφορία πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Και εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67. Χωρί ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 αποχές, απορρίπτεται. 70 το αρχικό κείμενο, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73. Χωριστή ψηφορία. Ονομαστική. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 74. Χωστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τίτλος με το 74 αρχικό κείμενο χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές και εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Έξι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 84. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 85. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 87. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Για το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Πέρασε. Ε, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 91. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά χερ εγκρίνεται 92 χωριστή ψηφορία ονομαστική πρώτο τμήμα ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98. Χωριστή ψηφορία ονομαστική. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Α, αποχές εγκρίνεται. 104. Πρώτο τμήμα Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουν. Πέρασε. Εγκρίνεται. 105 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 106. έξι. Χωριστή ψηφορία πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Εκατόν 8. Χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111. Αρχικό κείμενο. Χωριστή ψηφοφορία. Παντού με ονομαστική. Πρώτο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Mm-hmm. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 114. Χωριστή ψηφοφορία. Ονομαστική πρώτη μου. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουν. Πέρας. Εγκρίνεται. 119. Χωρίς τη ψηφορία πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία υπαρθμών. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσμα. Πέρασε. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Και τώρα προχωρούμε ε, στην επόμενη ψηφοφορία. Η 20η επέτειος της Ενευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον. Έχουμε την πρόταση ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτωται. Ήταν η πρόταση του ΕΝΕΦ. Και τώρα έχουμε το κοινό ψήφισμα από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Τροπολογία παριθμών 3 και προφορική τροπολογία πρέντα. Το κουμπί, το κουμπί του μικροφόνου. Για ξαναδοκιμάστε. Α, τώρα τα κατάφερα, επιτέλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρότασή μας λέει ότι στην τροπολογία 3 να διαγραφεί το τελευταίο κομμάτι εκεί που λέει ending in origin γιατί αυτό είχε ερμηνευθεί από τους ε, Βόσνιους ως εθνοκάθαρση και είναι απαράδεκτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει ένα κείμενο το οποίο λέει ότι θα πρέπει να γίνει εθνοκάθαρση βάρος των μουσουλμάνων στην Βοσνία Ριζεκοβίνη. Την προφορική τροπολογία υπάρχει κάποια ένσταση. deci Και τώρα Θα ψηφίσουμε αυτή την πρόταση ψηφίσματο. Υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Στέγκης. Πέρασε. Adoptat. Και εγκρίνεται. Και τώρα προχωρούμε στο 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. Πέντε νομιστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Ε, εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 6 καταπίπτει. 1 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος ψηφίζουμε τώρα με ονομαστική ψηφοφορία. Τώρα. Πέρας. Το ψήφισμα εγκρίνεται. Και προχωρούμε προς την ε, έκθεση Βαλέρο για τις εξαγωγές όπλων. Ένα. Χωριστή ψηφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5. Κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επτά. Κατά τμήματα. Πρώτο, πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οκτώ. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εννέα Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έντεκα Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ας γίνει έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος για το τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεκατέσσερα Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. υπέρ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεκαεννέα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά εποχές έλεγχος ηλεκτρονικός έλεγχος για την 20 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 26 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 ονομαστική ψηφοφορία Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 32. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 κατά τμήματα 5 τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συγγνώμη, εγκρίνεται το τρία, συγγνώμη. Ας κάνουμε έλεγχο, λέει και ο πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας γίνει έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 41. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 42 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 κατά τμήματα, τέσσερα τμήματα, ονομαστική ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54. Κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές ας γίνει έλεγχος για την 58 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 59 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται ετελογική σκέψη δέλτα δι λατινικό κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία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 εγκρίνεται. Προχωράμε λοιπόν, πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επιφυτικής ποικιλία. Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 2 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Νομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Ακόμα συνεχίζεται η ψηφοφορία. Τώρα περατούτε. Απορρίπτεται. Προχωράμε. Πάμε στο σημείο 4 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται.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 κατά άποχες εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Το επόμενο σημείο, η προστασία του Εθνικού Πάρκου Βιρούγκα στη Δημοκρατία του Κονγκό. 6 υπέρ. Κατά, άποχες, εγκρίνεται. Ένα υπέρ. Κατά, άποχες, εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Α γίνει έλεγχο, ηλεκτρονικό έλεγχο Για την τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο σας εύχομαι.